Uh, Καθίστε αγαπητοί φίλοι, λέει ο πρόεδρος. Στα πολωνικά. Α, ακούστε. Στις 2 Δεκεμβρίου διακόπησαν οι εργασίες μας, οι οποίες συνεχίζονται τώρα. Τα πρακτικά τη 13 η 11ης και 1 η Δεκεμβρίου